μάλυνση τη κατάσταση. Και επίση η δική μα χρηματοδότηση δεν μπορεί να πάει στα χέρια τρομοκρατών σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νοικοδόμηση αν δεν υπάρξει μια ισχυρή πολιτική διαδικασία πρώτα. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά συγκεκριμένων ατόμων και οντοτήτων, καθώς επίσης και απέναντι σε όλους τους αξιωματούχους εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την καταστολή κατά του Συριακού λαού. Όπως είπα και πριν από λίγο, η διένεξη αυτή στη Συρία, η σύγκρουση στη Συρία, αποτελεί πραγματικά ένα γεωπολιτικό αγώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι επικεφαλής διαδικασία για την προστασία τόσο των Συρίων όσο και των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειέ μα για το κοινό μα συμφέρον, συνεργαζόμενο με άλλου διεθνεί φορεί, με τη Ρωσία, την Τουρκία, τι Πολιτείες και άλλε χώρε. Και ελπίζω ότι θα έχω τη δυνατότητα να σα ενημερώσω για τις συζητήσει που θα έχω στην Ουάσιγκτον για το ζήτημα αυτό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ είπατε εκπρόσωπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Είπατε κι εσείς ότι βρίσκεται στο ένατο έτος του ο πόλεμος στη Συρία και πραγματικά ε, πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος. Στο τέλος φαίνεται από τις εξελίξεις ότι ο Ασάντ τελικά θα ενισχύσει τη, θέση του Ακόμη και οι τελευταίοι άμαχοι διαφεύγουν ως πρόσφυγες αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωπο αυτή τη στιγμή βρίσκονται διαρκώς εκτοπιζόμενοι, όχι απλά εκτοπισμένοι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Και για αυτόν τον σκοπό χρειάζεται να συνεχίσουμε τα αναπτυξιακά έργα στις ε, εμπόλεμες περιοχές. Περίπου το 60% των εκτοπιστέντων είναι παιδιά. Γι' αυτό και θέλω να κάνω έκκληση τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει τα παιδιά, τα σχολεία τους, μέσα στους καταβλισμούς των προσφύγων. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά, αλλά είναι απαραίτητα για, για το μέλλον των παιδιών, για να μην χάσουν τις ευκαιρίες τους. Βεβαίως ούτε αυτό αποτελεί φυσικά μια, μια μακροπρόθεσμη λύση. Αυτή τη στιγμή το πεπρωμένο της Ιντλίμπ εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας, Άγκυρας και Δαμασκού. Και σας Καλό να μου απαντήσετε. Ποιο θα είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί σωστά αναφερθήκατε στο ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ. Θεωρώ όμω ότι μια μακροπρόθεσμη λύση μπορεί να δοθεί ε, μόνο μέσα ε, από, τον, ε, από τα Ηνωμένα Έθνη. Αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω. Όμω θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει και έναν ισχυρότερο ρόλο όσον αφορά την επίτευξη Μακροπρόθεσμη λύση. Ευχαριστώ εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η κυρία Κάτι Πύρη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στη σημερινή συζήτηση για την κατάσταση ασφαλείας στη Συρία Δυστυχώ χαρακτηρίζεται από μια ε, τραγική ηρωνία. Γιατί η κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφάλεια στη Συρία. Δεν υπάρχει ασφάλεια για του εκατομμύρια αμάχου που ε, πρώτα εκτο, εκτοπίστηκαν στην περιφέρεια και τώρα βομβαρδίζονται στην Ιντλίπη. Υπάρχει μόνο καταστροφή, τραυματισμοί και θάνατος. Για εκείνους που νοσηλεύονταν στο, στα 56 νοσοκομεία που βομβαρδίστηκαν, στους, τους 300 που πέθαναν στους βομβαρδισμούς χωρίς τροφή, χωρίς στέγη. Για μια ακόμη φορά το Συριακό καθεστώς και οι υποστηρικτές του στη Ρωσία και στην, ε, στο Ιράν συνεχίζουν την τακτική τους, την απάνθρωπη, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές του ανθρωπισμού. Ελπίζω κάποια στιγμή ο Μπάσαρ Ασάντ να βρεθεί στην πόλη μου, στη Χάγη, ώστε τουλάχιστον να απονεμηθεί ένα μέρος της δικαιοσύνης για όλα όσα έχει διαπράξει εις βάρος ε, εκατομμυρίων Συρίων. Ευχαριστώ για το Ρινιού. Η κυρία Βάουτμαντς έχει το λόγο για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Μπορέλ, από το 2018 ξέρουμε ότι το Ιντλίμπ ε, ε, υφίσταται τεράστια πίεση από το καθεστώς ε, Ασάντ. Πέρυσι τον Οκτώβριο η Αμερική άφησε το Συριακό λαό στη μοίρα του και η Ευρώπη τα ίδια. Δεν κάνει τίποτα για τη δημοκρατική αντίσταση είναι ένας πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας δι' αντιπροσώπων. Εκατομμύρια είναι οι πρόσφυγες. Τα είπαμε όλοι. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, τι οφείλει να κάνει η Ευρώπη. Είναι πιο εύκολο φυσικά αυτό να το ρωτάς παρά να το απαντάς. Το κατανοώ πολύ, αλλά θα πρέπει να είναι ειλικρινής η Ευρώπη και να μην αφήσει την κατάσταση να εκφυλιστεί. Έχουμε τον Τραμπ εκεί να αποσύρεται και η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανασφαλής. Και αυτό που δεν μας βοηθάει είναι ε, το Συμβούλιο που είναι διχασμένο. Η Ιταλική κυβέρνηση τώρα επιζητεί προσέγγιση ε, με τον Ασάντ. Ε, εγώ δεν κατηγορώ τους Ιταλούς, κατηγορώ την Ευρώπη που δεν έχει μία φωνή. Η Ευρώπη θα βοηθήσει για τη βιώσιμη λύση μόνο όταν έχει μία ενιαία στρατηγική. Και πιέζει ο χρόνος. Και η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν λόγο να ε, χαλαρώσουν την πίεση στον Ασάτ. Θα πρέπει η Ευρώπη να φέρει ένα νέο σχέδιο για όλους. Και για μένα ο μοναδικός και ο πρώτος στόχος είναι η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός ε, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και τις γυναίκες και τα παιδιά εκεί. Ευχαριστώ ε, από την Ταυτότητα και Δημοκρατία, το λόγο έχει ο κύριος Μαριανή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εννιά χρόνια ε, φρίκης και η Ευρώπη συνεχίζει. Πολλά κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακραία στάση για το Συριακό. Είχαμε από τη μια το καλό, ε, του Αντάρτε, από την άλλη το κακό που ήταν η Συριακή κυβέρνηση και μετά ήρθε η πραγματικότητα. Σε λίγε εβδομάδε, τα φαβορή των Δυτικών εξουδετερώθηκαν από μια Ισλαμική φράξια γιατί ήταν πολύ μικρή αντιπροσώπευσή τους. Και στη συνέχεια έχουμε ε, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Γαλλίας, κατά των χριστιανών εκεί και αλλάζουν οι σημαίες ε, για να ε, φανούν αρεστοί πότε στον Ερντοάν, πότε στους Σαουδάραβες. Βλέπουμε λοιπόν τους τζιχαδιστές στο Χαλέπι. Η Γαλλία έθελε ότι φλούσε ως προς την ιδεολογία και την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκε με ε, μάλλον βρήκε, ε, ε, πιάσανε στην Μασαλία έναν υπεύθυνο της αντίστασης υποτίθεται με βίζα Εράσμους. Θα πρέπει τώρα, λέει στο Ιτλίπ, να προστατεύουμε τους τζιχαντιστές. Θυμίζω ότι είπε το Συμβούλιο Ασφαλείας τον περασμένο Ιούλιο. Το Ιτλίπ είναι αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτεροι δεξαμενοί ξέρουν μαχητών στον κόσμο. Ναι, να φροντίσουμε τους αμάχους, αλλά τους τρομοκράτες τι να τους κάνουμε. Στην Ευρώπη δεν τους θέλουμε. Άμα είναι ε, καλοί αντάρτες, γιατί δεν τους θέλει κανείς. Ή θα αφήσουμε την κυβέρνηση να κάνει ό,τι κάνουν οι κυβερνήσει στην επικράτειά τους, να ανακτήσει τον έλεγχο και να φέρει την ειρήνη εξολοθρεύοντας τους αντάρτες. Νόημαν, ένα λεπτό παρακαλώ, από τους πρασίνους. Μετά το Ιτλίπ μάλλον προς το Ιντλίπ ε, πήγανε όσοι δεν μπορούσαν να φύγουν από τη Συρία. Είναι εγκλωβισμένοι τρία εκατομμύρια σε ένα πόλεμο αντιπροσώπων και την πληρώνουν οι πιο αδύναμοι. Σχολεία, νοσοκομεία, ε, βομβαρδίζονται. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο Ιτλίπ είναι πραγματικά το δίκαιο όχι του ισχυρού αλλά του φρικτού. Βεβαίω θα πρέπει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πρέπει να κάνουμε ε, ό,τι μπορούμε. Πλήρη δημοκρατική ε, δράση, κυρώσει ε, και απέναντι στη Ρωσία και στην Τουρκία, στους υπευθύνους. Και φυσικά θα πρέπει να έχουμε ποσοστώσεις για τους πιο αδύναμους, που να τους υποδεχτούμε όσους μπορούν να βγουν από το ΕΤΛΥΠ δεν έχουμε συνολική λύση για τη Συρία, κύριε Μπορέλ. Προφανώ, κανεί δεν την έχει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά να κάνουμε τα μικρά βήματα που μπορούμε να τα κάνουμε με συνέπεια και να απαντήσουμε σε αυτή τη φρίκη στη Συρία, να αντιτάξουμε κάτι. Μια ελπίδα και ελπίζω ότι Δευτέρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να κάνετε ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, ε, Τζαμπάσκι, εξ ονόματο των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πατεκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα ένα ερώτημα το οποίο μας θέσατε. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το κάνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρετε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει από εσά. Αυτό είναι σαφές. Ουδής επίσης από τις κυβερνήσεις σας δεν πρόκειται να κάνει οτιδήποτε μέχρι να αρχίσετε να πουλάτε όπλα σε οδική Αραβία και εφόσον εθροτυφλείτε απέναντι στον Ερντογάν, άμα τους ε, αντιμετωπίζετε μόνο ως ε, ήπιους μετριοπαθείς Ισλαμιστές. Αν δεν τα αποδεχτείτε όλα αυτά, απλώς θα αναλωνόσαστε σε συζητήσεις σαν τη σημερινή. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι ο μετριοπαθής αυτός Ισλαμισμός κόβει κεφάλια χριστιανών όμως. και αυτοί που χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις σας είναι πραγματικά προδότες, πολεμιστές και θα συνειδητοποιήσετε ότι εσείς τίποτα απολύτως δεν μπορείτε να κάνετε. Από τελικού, ε, παρακαλώ, κύριος Γεωργίου. Έχετε το λόγο. Για ένα λεπτό. Κύριε Μπορέλ, οι πόντοι, οι πιλάτι δεν μας χρειάζονται. Καθώς η τραγωδία στη Συρία είναι πλέον απερίγραπτη επειδή κάθε νέα της πτυχή είναι και πιο ντροπιαστική. Το τελευταίο επεισόδιο διαδραματίζεται στο Ιντλίπ, εκεί όπου 700 Σύριοι φοιτητέ έχουν απαχθεί από τρομοκρατικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία, άλλοι ναρκώνονται και άλλοι φανατίζονται και ρίχνονται στην πολεμική κρεατομηχανή. Έναν εκατομμύριο άνθρωποι έχουν προσθεθεί στις προσφυγικές ροές. Η ζώνη ασφαλείας που θα δημιουργούσε ο ταγίπ ερντογάν ο ανηλεής Ερτογάν έχει ανοίξει τις πύλες της κολάσεως. ακούτε τι συμβαίνει. δεν μιλάμε για ψυχρούς αριθμούς μιλούμε για ανθρώπους μιλάμε για μικρά παιδιά τα οποία έχουν όνειρα και ψυχή ή αυτά δεν λογαριάζονται. στη συρία κρίνεται τον Boeing της ευρώπης στην ανατολική μεσόγειο κρίνεται το κύρος της ανθρωπότητας τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη ή τα αφήνουμε σε διαβολικά μυαλά ή στι διαβολικέ δαιμονικές δίθεν συμφωνίε του αιώνα. Ιζαμπέλ Σάντος έχει το λόγο για ένα λεπτό εξ των Σαλιστών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε. Βλέπουμε ότι περίπου 600 Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα στους τελευταίους μήνες. Μα νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική δεχτής κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Συρία. Και έχουμε μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση επίσης. Η χώρα έχει ήδη καταστραφεί μετά από τον εναετή αυτόν πόλεμο και όσοι έχουν επιβιώσει βιώνουν απερίγραπτη οδύνη. Πάρα πολλέ επιθέσει στρατιωτικέ στον άμαχο πληθυσμό, καθώ επίση και στι υποδομέ του άμαχο πληθυσμού ακόμα και στους καταβλισμούς εκείνους που έχουν δημιουργηθεί για τους αμάχους, οι οποίοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες στέγασης, καθώς επίσης και σε κάποιες πολύ πρωταρχικέ σημαντικέ υπηρεσίε. Θα πρέπει λοιπόν τον άμαχο αυτό πληθυσμό να συνεχίσουμε να τον βοηθάμε, λαμβάνοντα όμω τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη πλέον συμφωνία, η οποία να συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Αρμοστία για τους πρόσφυγες κάνει έκκληση για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, όπου θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου οι ανθρωπιστικές ομάδες να μπορούν να φτάσουν στον άμαχο πληθυσμό. Πραγματικά η ανταπόκριση στην έκκληση αυτή ποια ακριβώς ήταν, μπορείτε να μα πείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρετχεν για ένα λεπτό. Vielen Dank. Ευχαριστώ. Από το Φεβρουάριο του 2019, το αναφέρατε κύριε Μπορέλ, η σύγκρουση οξύνεται. Υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι και από το Σεπτέμβριο του 2019, συνάδελφοι, ε, σκεφτείτε το, το Ιντλιπ και η περιοχή ε, βαμβαρδίζει σχεδόν καθημερινά από τον Ασάντ με την υποστήριξη της ρωσικής αεροπορίας. Από το, την Παρασκευή το βράδυ η Τουρκία έστειλε πάνω από 600 πολεμικά αεροσκάφη πάνω από τα κοινά σύνορα. Ε, εκφράζονται φόβοι για ε, περαιτέρω όξυνση τη σύγκρουση μεταξύ Συρίας και Τουρκία. Από το Δεκέμβριο πάνω από 500.000 άνθρωποι είναι πρόσφυγε, 80% γυναίκε και παιδιά. Αυτό αυτός ο εκτοπισμό είναι ένα από του μεγαλύτερου από την αρχή τη ε, σύγκρουση το 2011. Συνεχίζεται η σύγκρουση λοιπόν και ε, στη διάρκεια αυτής έχουν ε, χάσει τη ζωή τους πάνω από 400.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 220.000 παιδιά και εμεί οι Ευρωπαίοι απλά κοιτούμε ω παρατηρητέ. Πρέπει επιτέλου να βρεθεί μια πολιτική λύση, πρέπει να πετηθεί μια πολιτική λύση. Το είπε και ο κύριο ε, Μπορέλ. Ναι, αλλά τι σημαίνει συγκεκριμένα αυτό ε, ανόκρανη του ΟΗΕ. Τι ακριβώς, ε, ποιο ακριβώς είναι το όραμά μα για αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε ηθική υποχρέωση να έχουμε και ένα συγκεκριμένο όραμα για την περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβάν Ντάβιντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το βασικό πρόβλημα στην ε, Συρία είναι η διαπραγματευτική ισχύ τη Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη και διεφθαρμένη, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον πρώτο λόγο έχουν οι πολυεθνικέ. και αυτέ δεν έχουν κάνει πραγματικέ επενδύσει ποτέ στην Τουρκία, ώστε να έχει κάποιο βάρο ειδικό ο λόγο του. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε αυτή την αποδυναμωμένη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να επιβάλλει και κυρώσει στην Τουρκία. Αντιθέτω την βοήθησε να επιβάλλει η Τουρκία δηλαδή κυρώσεις εναντίον της Συρίας. Βεβαίως ακυρώθηκαν ορισμένες πληρωμές στην Τουρκία. Ε, από την άλλη πλευρά ε, χορηγήθηκαν όμως ε, από άλλες πλευρές χρήματα στην Τουρκία ακριβώς γιατί ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση η φύλαξη των συνόρων της. Γι' αυτό και η Τουρκία έχει ενισχυμένη θέση. Παρά το γεγονό ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο Κούρδου και Χριστιανού. Και παρά το γεγονό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον, δεν είναι σε θέση να φροντίσει ούτε καν τον ίδιο τον εαυτό της και δεν απαγορεύει στην ε, Τουρκία ούτε καν να προχωρά σε παράνομε εξορίξει φυσικού αερίου στη Βόρεια Κύπρο. Κυρία Κακό έχει το λόγο. Από το 2011 400.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε λοιπόν για μια σύγκρουση που διονύζεται. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί επιγόντω μια λύση. Η οδύνη του Συριακού λαού, καθώ επίση και ο κίνδυνο να έχουμε μια μακροχρόνια στάθεια, εφίσταται για πάρα πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν δώσει πάνω από 70 δισεκατομμύρια σε βοήθεια και το Συμβούλιο έχει επιβάλει και κυρώσει. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά δεν αρκούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ επίση και άλλοι διεθνεί φορεί θα, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να σταματήσει η διένεξη αυτή και να βρεθεί τελικά μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει στην ειρήνη. Η επιρροή όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί αν δεν είναι σε θέση να μιλάει με μια ενιαία φωνή τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση όσο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πρέπει αυτή τη στιγμή να δείξουμε ρεαλισμό καθώς επίσης και διπλωματική αποφασιστικότητα. Στο πράξουμε λοιπόν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νικολάη Βίλουμσεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η επανάσταση στη Συρία ξεκίνησε ως λαϊκή εξέγερση εναντίον της βίαιης δικτατορίας. Η εξέγερση αυτή βεβαίως αντιμετωπίστηκε με ε, ε, τεράστια καταστολή ε, και δυστυχώς η Ευρώπη δεν κατάφερε να υποστηρίξει την εξέγερση αυτή. Τώρα η Συρία έχει, έχει μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων όλων των μεγάλων δυνάμεων στον κόσμο. Ο πρόεδρος ε, Ερντογάν αξιοποιεί τις ε, μιλιταριστικές του πολιτοφυλακές για να, ε, δημιουργεί, για να προχωρά σε καθαρίσεις επί Συριακού εδάφους, ενώ ο Πούτιν χρησιμοποιεί τη δική του στρατιωτική δύναμη, συνεχίζοντας κανονικά χωρίς καμία επίπτωση τις, ε, τις παραβιάσεις του διεθνούς ε, δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην, ε, στον αγώνα και κατά του Νταές και κατά του καθεστώτος του Ασάντ. Πρέπει επιτέλους να επιβάλλουμε κυρώσεις έως ότου σταματήσουν οι παραβιάσεις, οι εισβολές και έως ότου ο ΟΗΕ μπορέσει να στείλει ηρευτική δύναμη στην βορειοανατολική Συρία ώστε να εξασφαλιστεί από την εκαθάριση ο Συριακός λαός. Αυτό πρέπει να είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Μπορέλ. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει μπλε κάρτα για εσάς. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Αποδέχεστε την μπλε κάρτα. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον τελευταίο μιλητή. Ποιο είναι ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Σαουδική Αραβία, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είναι σταθεροποιητικός συμφωνείτε ότι είναι πόλεμος δι' αντιπροσώπων, αλλά και με παρέμβαση αυτών όλων των δυνάμεων που έχουν ε, οπλίσει ε, τους αντάρτες ε, για να ρίξουν τον Άσαντ. Και είναι ανοησίες αυτά που λέγονται ότι οι Κούρδοι έχουν πρόβλημα με τον Άσαντ. Με την Τουρκία έχουν πρόβλημα οι Κούρδοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα χέρια της αιματοβαμμένα. Απάντηση. Φυσικά υπάρχει γεωπολιτικό ενδιαφέρον και συμφέροντα για τη Συρία, αλλά υπήρχε και ειρηνική διαδήλωση από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στη Συρία που ζητούσαν ελευθερία, δημοκρατία. Και αυτή η κραυγή λαού πατάχθηκε ε, δρυμύτατα με καταστολή του καθεστώτος του Ασάντ, εμεί θα πρέπει να κάνουμε, να είμαστε στο πλευρό των Κούρδων και των φιλοδημοκρατικών δυνάμεων που αγωνίζονται για τη δημοκρατία και την ειρήνη. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα και στη Συρία και στη Μέση Ανατολή ολόκληρη. Ευχαριστώ, κύριο Πίτσουλα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εννιά χρόνια, όπως ακούσαμε, ακού, ε, διαρκεί ο πόλεμος αυτός ε, στην Συρία και είχαμε κλιμάκωση το τελευταίο αυτό διάστημα και οξύνεται ιδιαίτερη ανθρωπιστική κατάσταση όπως και στην Ιεμένη. Ας μην ξεχνάμε ότι 400 περίπου χιλιάδε άτομα ήδη από το Δεκέμβριο έχουν εκτοπιστεί και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το 80% των προσφύγων αυτών ήδη ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, γυναίκες και παιδιά. Υπάρχουν πολλοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί που, ε, αναγκάστηκαν να σταματήσουν τι επιχειρήσει του. Ένα τέταρτο παιδιών δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στο σχολείο. 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη. Και η ανθρωπιστική αυτή κρίση επιδεινώνεται και από τι μετρολογικέ συνθήκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ω παράγοντας που προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα θα πρέπει να αναλάβει όχι πλέον θεωρητικό αλλά δραστήριο ρόλο που θα προτείνει λύσει. Θα πρέπει να εντείνουμε τι συζητήσει μεταξύ των συμβαλωμένων μερών αλλά και να καταφέρουμε να προσφέρουμε μια πολυμερή πλατφόρμα για την επίλυση, την πραγματική επίλυση τη κρίση. Α ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη πρόσφατη διάσκεψη τη Βρυξέλλε που έδωσε μια, κάποια αποτελέσματα για τη Λιβύη. Ο κύριο Γκλουξμάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πατεκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, α κοιτάξετε όλοι τα βίντεο που έχουν βγάλει στα ε, κοινωνικά μέσα τις τελευταίες μέρες οι ε, στρατιώτες του Μπασάρ. Ε, ξεθάβουν πτώματα, γελάνε, βασανίζουν τον κόσμο. Αυτό είναι ε, σαν να φτύνουν τον κόσμο. Ε, οι Ρώσοι μαζί με τους ε, Σύρους θερίζουν ε, νοσοκομεία, σχολιά, φούρνους κλπ. και τους αφήνουμε όπως αφήνουμε εδώ και 9 χρόνια. Ακούω ορισμένους εδώ να υπερασπίζονται το καθεστώς και να ζητούν την εξολόθρευση των ανταρτών. Να σας πω ότι ντρέπομαι και νιώθω αποτροπιασμό. Κύριε Πατεκπρόσωπε, να μην υποχωρήσετε ποτέ σε αυτές τις ειρήνε εξομάλυνσης με το καθεστώς του Ασάντ. Να μην ξεχνάμε ποιοι είναι οι φίτες και τα θύματα. Και ο Μπασάρ, ε, η θέση του είναι στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και πουθενά άλλου. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, προχωρούμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ, όπου έχουν ζητήσει το λόγο οκτώ συνάδελφοι. Ε, σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας ένα λεπτό έκαστος. Ο κύριος Μπασέσκου πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. σε σχέση με τη Συρία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διέλθει διάφορα στάδια, διάφορες φάσεις. Στην αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε το κεφάλι του Πασάρ Ελασάντ επί πινακίου. Τα τελευταία χρόνια λέμε ότι δεν θέλουμε το κεφάλι του, θέλουμε όμως να κριθεί. Θέλουμε εκλογές στη Συρία. Αυτό είναι έλλειψη συνέπειας και δίστασα από την αρχή, διστάσαμε θα έλεγα. Διστάσαμε όσον αφορά την παρέμβαση, δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε τους Γάλλους από παρέμβαση και τώρα διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση στη Συρία. Η Συρία θα παραμείνει υπό ρωσικό έλεγχο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παραπονεθήκαμε λέγοντας ότι η Τουρκία εισβάλλει στη Βόρεια Συρία. Οποιαδήποτε χώρα θα το έκανε αυτό για να προστατεύσει τα σύνορά της. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο δεν κατανοούμε ότι το να μπορούμε να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων σημαίνει κάποια συμμετοχή. Συνέχεια θα καταγγέλουμε την καταστροφή στη Συρία. Είτε θα παρέμβουμε ή θα αφήσουμε τους Γάλλους να παρέμβουν και αν είναι να παρέμβουμε δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε ευθύνε για αυτά που συμβαίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος συνάδελφος είναι ο κ. Ρόι Τέβες. Ε, για ένα λεπτό. Α δώσουμε τη δυνατότητα σε όλου που θέλουν να μιλήσουν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον είπα το εκπρόσωπο για την έκκληση που κάνω όσον αφορά την Συρία. Δεν θα το επαναλάβω. Υπάρχουν επιθέσεις εναντίον των αμάχων, υπάρχουν ε, οι νεκροί, οι φρικαλαιότητες, τα είπαν πολλοί συνάδελφοι εδώ. Εννοείται ότι όλα αυτά τα καταδικάζουμε. Επιμένουμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά είναι αλήθεια επίσης ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην πράξη αποτελεσματικά. Στην περίπτωση της Λιβύης η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε να δηλώσει εμπάργο όπλων και το εκπρόσωπος φρόντισε ώστε να είμαστε εμείς εκείνοι που θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του εμπάργου. Βέβαια, το Συριακό καθεστώς διαθέτει όπλα. Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε είναι κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε εμπάργο όπλων στο καθεστώς του Σαραλασάντ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Μίλλερ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς τώρα παρακολουθούμε πάλι μια τραγική κατάσταση. Πρώτα απ' όλα μια ανθρωπιστική κρίση με εκατομμύρια προσφύγων οι οποίοι φεύγουν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και πηγαίνουν στην Τουρκία ή είναι στα σύνορα με την Τουρκία. Έπειτα έχουμε την εισβολή την τουρκική στη Συρία που βέβαια δεν βοηθάει να αποφύγουμε τον πόλεμο και τρίτον παρακολουθούμε τον τουρκικό στρατό να πολεμά την αλκαΐδα. Λοιπόν, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πια θα μπορούσε να διαπραγματευτεί και να πιέσει την Τουρκία εδώ που βρισκόμαστε. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να αντιταθούμε στην δίωξη των Κούρδων και να αντιταθούμε στις φρικαλαιότητες των τζιχαντιστών αλλά και της Τουρκίας κατά των Κούρδων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαυρίδη είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να το ξεκαθαρίσω κύριε Μπορέλ. Δεν είμαι καθόλου θαυμαστής του καθεστώτος Άσαντ, του οποίου τα χέρια είναι βουτυγμένα στο αίμα. Αλλά ακούγοντα σήμερα κάποιε από τις απόψει νομίζω υπάρχει μια σύγχυση. Θεωρούσα μέχρι τώρα ότι είχαμε ομόφωνη απόφαση ότι ο στόχος μας και της δύσης του πολιτισμένου κόσμου είναι η εξουδετερώση του ισλαμικού κράτους και των τζιχαντιστών. αν άλλαξε κάποιοι να το πουν δημόσια. επομένως το ερώτημα είναι ποιος χρηματοδοτεί τους τζιχαντιστές ποιος στέλνει στρατεύματα για να συνεχίσουν να κάνουν τις σφαγές τους ποιος τους χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια έχει όνομα αυτός είναι ο νεοσουλτάνος στην άγκυρα και το όνομα αυτού είναι ρατζίπ Ερτοάν. αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας και όσοι το λέμε δεν είναι γιατί συγχωράμε τα εγκλήματα του άσαντ είναι γιατί έχουμε την τόλμη να λέμε την αλήθεια γιατί πιστεύουμε στις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κέμπα έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε. Συμφωνώ με αυτά που είπατε στην αρχή, ότι δηλαδή στη Συρία αλλά και στις γείτονες χώρες έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωπιστική καταστροφή. Κάπου 10.000 ε, περίπου βρίσκονται στο Λίβανο, για παράδειγμα, που χρειάζονται βοήθεια αμέσως. Η δικιά μου χώρα εμπλέκεται και πέρα από τη συνεισφορά μας στους ευρωπαϊκούς στόχους έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε περισσότερα κονδύλια στην ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο, τη Συρία κλπ. και την Ιορδανία. Αυτό που λέτε για επενδύσεις, για κονδύλια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου είναι ο μεγαλύτερος όμως έχουμε και πληροφορίες ότι από το 1,5 εκατομμύριο χριστιανούς κάπου 200.000 έχουν μείνει. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν είναι τραγική. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, τις αποστολικές αρχές που βοηθούν τα παιδιά που προσφέρουν ιατρική αρρωγή. Είναι μια έκκληση που κάνω σε ολόκληρο το κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σάντρα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή που ε, μιλάμε, ο στρατός και οι σύμμαχοι προελάβουν ε, και ανακτούν τον έλεγχο κατεχόμενων ε, από τρομοκρατικές ομάδες περιοχών. Και η σημερινή συζήτηση έχει σχέση με ένα στρατιωτικό κομβόι και με επιθέσεις από πυράβλους από το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθούμε τον έλεγχο των φυσικών πόρων ε, της Συρίας ε, και να αφισβητήσουμε την νομιμοποίηση των Συριακών αρχών γιατί πρόκειται για μια γεωστρατηγική περιοχή. Αυτό είναι ο στόχος, αυτά είναι τα συμφέροντα της Realpolitik τελικά και αυτό έρχεται σε βάρος με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουμε να το καταδικάσουμε το ε, ζήτημα αυτό, η ε, επίλυση της σύγκρουσης, ε, σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούμε ε, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα. Και το διεθνές δίκαιο επίσης πρέπει να γίνει σεβαστό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Συριακός στρατός προχωράει εναντί της Τουρκίας και των τζιχαντιστών που στηρίζουν η ΙΠΑ στην περιοχή του Ιτλίμπ. Η Συριακή κυβέρνηση αποκαθιστά τα σύνορά της και βρίσκει πάρα πολλά αμερικανικά όπλα ως το κάνουν οι τζιχαντιστές. Η επαρχία του Ιντλίπ ε, κυριαρχείται από τις διάφορες ε, ομάδες της ε, Αλκάιντα. Αυτοί οι τζιχαντιστές εκπαιδευόταν και βοηθόταν από μιλητή από τη Βρετανία, την Τουρκία, τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτω από το πρόγραμμα Σίκαμορ του Ομπάμα και κατέληξε η όλη πολιτική σε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους ε, που δεν χρειαζόταν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ζητά πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια στην επαρχία του Ιντλίπ χωρίς περιορισμούς. Ή επιβάλλουμε ε, κυρώσεις που δημιουργούν πολλές κακουχίες στο Συριακό λαό. Γιατί δεν τους παίρνουμε πίσω, τους, τους θέλουμε όμως οι Dziękuję. Panie pośle, głos pani poseł Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, κυρία Ντάνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αναμφισβήτητα ο Συριακός λαός ε, υπέφερε επί 9 χρόνια και παραπάνω. Αλλά γιατί συνέβη αυτό. Διότι η δυσαρέσκεια του λαού κατά της κυβερνήσεως Ασάντ αρπάχτηκε από διεθνείς φορείς που προσπάθησαν να πετύχουν ανατροπή του καθεστώτος και από τη ΣΥΠΑ και κάποια κάτι μέσα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τη υποστήριξη αυτών πέρασαν μέσω Τουρκία οι τσιχαντιστέ αυτή τη χώρα. Μετά από 10 χρόνια δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση που ανέκτησε τον έλεγχο. Και όπω ανέκτησε τον έλεγχο, ε, ρύθμισε την κατάσταση με το λαό. Κάποιοι συμφώνησαν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, κάποιοι άλλοι διαφώνησαν και πήγαν στο Ιντλίμπ. Αυτό ήταν επόμενο. Είναι ηρωνικό όταν μιλάμε για του ξένου μαχητέ, που ήρθαν από δικέ μα χώρε και δεν του δεχόμαστε να επιστρέψουν, αλλά περιμένουμε οι Σύριοι να αντιμετωπίσουν το θέμα, δεν είναι κατανοητό. Θα πρέπει να σταματήσουμε τι κυρώσει, να καθίσουμε με τη Συριακή κυβέρνηση και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη σε αυτή τη χώρα και να υπομισθούμε τι ευθύνε για το ρόλο τη Ευρώπη σε αυτή την καταστροφή και να παραδεχτούμε το ρόλο τη Συριακή κυβέρνηση που σταμάτησε ε, του τζιχαντιστέ και την άνοδο του ISIS. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο. Αντιπρόεδρος και τους Εκπρόσωπος, ο κύριος Γιαζέπ Μπορέλ έχει το λόγο. Ο κύριος Μπορέλ, Μπορέλ Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλες και όλους ε, τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Και δεν μπορώ να πω παρά ότι και κατανοώ και συμμερίζομαι την απογοήτευση πολλών όπως εκφράστηκε στις παρεμβάσεις διότι η κρίση στη Συρία ε, έχει δείξει ότι ήταν αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι και αν λέμε πρέπει, πρέπει, πρέπει να κάνουν αυτό, να κάνουν το άλλο. They should, faut, ε, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε όποια γλώσσα και αν το πούμε, με τι ε, δυνατότητα επιρροής, με τι ισχύ, με τι μόχληση μπορούμε να επηρεάσουμε. Πολλά χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Και τελικά υπήρξε στρατιωτική λύση στη Συρία. Ή, τέλος πάντων, αυτό βλέπουμε. Και από ποιον? Από αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική ισχύ. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση όμως η παντων αυτο βλεπουμε και απο ποιον απο αυτους οι οποιοι μπορουν να χρησιμοποιησουν Ένωση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να, να απευθύνουμε έκκληση σε όλους. Να τερματίσουν τις επιθέσεις σε βάρος του άμαχου πληθυσμού να πάψουν να εμποδίζουν ε, την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να σεβαστούν τους κανόνες και τις υποχρεώσεις ε, που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, να προστατεύσουν τους αμάχους. Ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι διακηρύξεις αρχών αλλά δεν έχουμε δύναμη εξαναγκασμού που να μπορούμε να επιβάλλουμε τελικά αυτά όσα ζητούμε. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία γίνονται στη Συρία είναι ένα μεγάλο μάθημα για την Ευρώπη, για αυτό το γεωπολιτικό πρωταγωνιστή που θέλουμε να γίνουμε. Αν θέλουμε να γίνουμε ουσιαστικά και αν θέλουμε θα πρέπει να προβούμε στι απαραίτητε ενέργειες και να έχουμε στη θέση μα και τα απαραίτητα μέσα. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε τέτοιε κοινοβουλευτικέ συνεδριάσει και θα συνεχίσουμε να λέμε πρέπει, πρέπει, πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Τώρα, συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Αυτό είναι ο τίτλος. Θέλω να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία Cards ή να κάνετε μια ερώτηση στα πλαίσια της διαδικασίας της μπλε κάρτας, μπορείτε και ηλεκτρονικά αλλά και διαντάσσεω χειρός να ζητήσετε το λόγο. Ο πρώτος θα πάρει το λόγο είναι ο συντάκτης της ερώτησης, πρόεδρος της Επιτροπής ε, ΔΕΒΕ, ο κύριος Τομπέ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ολοκληρωμένη αυτή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική είναι μια ευκαιρία για καλύτερες σχέσεις της Αφρικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρέπει να υποσχεθούμε ένα τον άλλον ότι προσπαθούμε να πάμε μπροστά με καλές προθέσεις και με συγκεκριμένες δράσεις. Ας φροντίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στις δράσεις και να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο. Μια νέα στρατηγική πρέπει να αναγνωρίζει τις δυνατότητες που έχει Αφρική. Υπάρχει ενδιαφέρον στρατηγικό για την Αφρική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζουμε τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για την Αφρική. Για να πετύχει όμως η στρατηγική μας για την Αφρική πιστεύω ότι χρειάζονται τα Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλουμε και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να χρησιμοποιήσουμε μια συνολική στρατηγική με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Δεύτερον, χρειάζεται συνειδητοποίηση για το τι μπορούμε να κερδίσουμε αν πετύχουμε την ενίσχυση τις σχέσεις μας με την Αφρική και τι διακυδεύεται αν δεν τα καταφέρουμε. Και τρίτον, πρέπει να προσδιορίσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ώστε να συντονίζει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις χώρες μέλη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά, πολλές ευκαιρίες, αμοιβαία εποφελής, ανάπτυξη, απασχόληση, εμπόριο. Υπάρχουν όμως και προκλήσεις, κλιματική αλλαγή, ένδια, ε, συγκρούσεις, και μετανάστευση. Η μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη που διαπιστώνουμε στην Αφρική σημαίνει ότι θα συνεχίσει αυτή η αύξηση και όσον αφορά την αγορά εργασίας. Σε λίγο εκεί θα είναι οι νέοι, στην Αφρική. Οι συγκρούσεις όμως δυστυχώς υπάρχουν και υπάρχουν εκεί που υπάρχει ένδια και υψηλά επίπεδα ανεργίας. Οπότε εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης έχω υποβάλει διάφορες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτον λοιπόν, πώς η στρατηγική αυτή θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και το στόχου της, ε, <clears throat> στόχους μας όσον αφορά την καταπολέμηση της ένδυας. Δεύτερον, πώς η νέα στρατηγική θα συνεισφέρει στην ενίσχυση και στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των ανισοτήτων κλπ. Τρίτον, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι θα συμμετέχουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών, στον σχεδιασμό της στρατηγικής αυτής. Τέταρτον, επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τον κίνδυνο επικαλύψεων. Μιλάμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι Αφρικανοί εννοείται ότι αποτελούν προτερότητα. Ε, μιλάμε επίσης για το μέλλον των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα διασφαλίσει συνέπεια και πώς θα αποφύγει τον κίνδυνο ε, στρατηγικών ε, που θα επικαλύπτονται μεταξύ τους. Και τέλος, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αναπτυξιακή πολιτική και η πολιτική συνοχής βρίσκεται εγγεγραμμένη στις πολιτικές μας, στις συνθήκες μας και πρέπει να τα καταφέρουμε. Γι' αυτό θέλω να ξέρω πώς θα διασφαλίσετε ότι θα συμπεριλάβετε στην, στο σχεδιασμό της στρατηγικής την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Ανάπτυξη και εγώ προσβλέπουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία. Α ξεκινήσουμε τη δουλειά μαζί. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Γιούτα Ουρπιλάινεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε στη συζήτηση ενός πραγματικού σταθμού, ενός ορόσημου στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρική. Αυτό είναι η νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αφρική. Είχα δεσμευτεί και στη διάρκεια τη ακρόασή μου ότι θα κάνω πάντα δυνατό για την ενίσχυση και την εμβάθυνση τη συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε σήμερα αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Δεν υπάρχει τίποτα καταλληλότερο για την πρώτη μου παρέμβαση ενώπιόν σας από μια συζήτηση για τη σχέση μας με την Αφρικανική Ήπειρο. Εκτιμώ ιδιαίτερα την εμπειρία της γνώσης, ε, της απόψης σας και θεωρώ ότι θα είναι σημαντικές για αυτό το ζήτημα. Στη ε, πρώτη μας ε, επίσκεψη εκτός Ευρώπης, η πρόεδρος Φοντρελάν και εμείς πήγαμε στην Αφρική και είδαμε μια νέα Ήπειρο ε, αισιόδοξη, γεμάτη δυναμικό ελκυστικό τόπο για τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές. Είναι ένας εταίρος ε, που αξίζει να είμαστε θετικά ε, δεσμευμένοι απέναντί του. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος για αλλαγή ε, στο πλαίσιο της συμμαχίας, για επενδύσεις σε θέσεις εργασίας. Έχουμε τη στήριξη του σχέδιου εξωτερικού, εξωτερικού σχέδιου επενδύσεων και έχουμε επίσης σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απτή πρόοδο και τώρα μπορούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και να προχωρήσουμε περί περαιτέρω και να ανοίξει πια ένα νέο κεφάλαιο που θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας. Για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτή η στρατηγική θα στηρίζει το δυναμικό της Αφρικής, τις προσπάθειες για την πολιτική οικονομική διακυβέρνηση και θα προωθεί την ειρήνη και την αντοχή την ανθεκτικότητα. Η στρατηγική που θα την κάνουν κτήμα τους οι Αφρικανοί. Επίσης θα τοποθετήσει την Ευρώπη σε μια καλύτερη θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο με βάση και τους στόχους αυτής της Γεωπολιτικής Επιτροπής και τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες. Ετέθησαν ήδη το 2017 και παραμένουν και σήμερα οι ίδιες. Ε, η προσέγγιση μας δεν είναι να αλλάξουμε κατεύθυνση, να αλλάξουμε πορεία, αλλά να ανεβάσουμε ταχύτητα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αυτή η στρατηγική και αυτό θα εξασφαλιστεί και από τις την ε, ε, άμεση σχέση με του στόχου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, του στόχου ε, για την ε, κλιματική αλλαγή τη Μόνα των Παρισίων, την συνολική μα στρατηγική, καθώ και την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη ε, και το θεματολόγιο 2063 της Αφρικανικής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την υπηρετική ολοκλήρωση, την οικονομική ολοκλήρωση, την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση μετανάστευση, επίση ε, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Θα εστιάσουμε και σε άλλου τομεί όμω, την ψηφιοποίηση, την ισότητα των φύλων, που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρί στέρη διακυβέρνηση και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όμω δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε χωρί σεβασμό στο κράτο δικαίου και τη δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα ε, στου τομεί αυτού παράλληλα με την ε, μάχη που θα δώσουμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι θέλουμε να συνεργαστούμε και με του Αφρικανούς εταίρου μας στο πλαίσιο ενό πολυμερού συστήματο βάση κανόνων, το οποίο τίθεται όλο και περισσότερο από αφισβήτηση στις μέρες μας. Μια βασική προτεραιότητα στην θητεία μου θα είναι να εξασφαλίσω ότι η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα υποστηρίζει τη δύναμη που αντιπροσωπεύει η νεολαία. Οι νέοι και οι νέε πρέπει να κάνουν κτήμα του αυτή τη στρατηγική. Έχουμε ένα νέο φιλόδοξο πλαίσιο. Ήδη έχει ξεκινήσει η εργασία μας από αυτού και σε πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο και στο μεταξύ συνεχίζουμε να αφουγκραζόμαστε και προσπαθούμε να υπάρξει οικειοποίηση, βιοποίηση αυτή της στρατηγικής από εσάς τους ίδιους αλλά και από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Το ίδιο και από τους Αφρικανούς μας εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των νέων. θα γίνει μια συνάντηση στις 27 ε, Φεβρουαρίου στην Αιθιοπία μεταξύ των ε, δύο πλευρών και η Υπουργική Διάσκεψη το Μάιο. Και οι δύο αυτές εκδηλώσει αποτελούν σημαντικέ ευκαιρίε για να έχουμε διάλογο με του Αφρικανού μα εταίρου. Προτίθεμαι επίση να μεταβώ το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στην Αφρική για να έχω διαβουλεύσεις, όσο δυνατόν ευρύτερε διαβουλεύσεις. Η πρόταση για τη νέα στρατηγική θα είναι στην μέση διάταξη των των επιτρόπων στις αρχές Μαρτίου προς έγκριση και αυτό θα σηματοδοτεί στην αρχή πιο συγκεκριμένης δουλειάς μαζί με τους ε, βασικούς ε, ενδιαφερομένους φορείς. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και κυρίως το να ακούσω τις δικές σας απόψεις, να ακούσω εσείς τι θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Εκ μέρου του ΕΛΚ, Χίντεργαρντ Πέντελε, έχετε το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε. Πραγματικά ξεκινά μια νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική, γιατί ε, η σημερινή επιτροπή έχει θεωρήσει αυτόν μια γεωπολιτική επιτροπή και πραγματικά υπάρχουν κατεπήγοντα προβλήματα. Κλίμα, μετανάστευση. Θα πρέπει να ανανεωθεί η Συμφωνία Κοτονού. Έχουμε και το Πράσινο Σύμφωνο Αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς ε, η ψηφιοποίηση και όλα αυτά είναι νέα ε, στοιχεία, είναι νέα δυνατότητες που πρέπει να καταλευθούμε στο πλαίσιο αυτής της νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής και για μένα είναι σημαντικό ε, να αξιοποιήσουμε όλη την εργαλειοθήκη με συνεκτικό τρόπο που έχουμε στη διάθεσή μας και επίσης να διδαχθούμε από το παρελθόν, από αυτό σημαίνει να εστιάσουμε πρώτα απ' όλα στις δίκαιες εμπορικές σχέσεις και στην δημιουργία εισοδήματος, σε δημιουργίες εκπαίδευση στην Αφρική Δημοκρατία και πρόσφυγη κράτους δικαίου. Ε, να έχουμε καλύτερες διοικητικές δομές, ε, προστασία γυναικών ε, και κοριτσιών. Και επίσης να παρέχουμε την βοήθεια πιο πολύ επιτόπου στοχευμένα. Θέλουμε να έχουμε εξασφαλισμένο το μέλλον και τις δυνατότητες για όλους τους Αφρικανούς, γυναίκες και άντρες στη χώρα τους. Ε, και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς Αφρικής έχουμε ευθύνη να έχουμε μια πραγματική εταιρική σχέση που θα είναι υποφελής και για τις δύο πλευρές. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ε, με την πρόταση που έκανε ε, για μια επίτροπο, για έναν την Αφρική, νομίζω δείχνει πόσο μεγάλη προτεραιότητα δίνουμε εμείς ως ΕΛΚ στην Αφρική και θέλουμε να χαιρετήσουμε την προσήλωσή σας και ελπίζουμε σε αυτή τη θητεία να έχουμε δημιουργήσει νέα θεμέλια για μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική της Ένωσης με την Αφρική. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ευχαριστούμε εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ούντο Μπούλμαν για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπα, αξιότιμοι συνάδελφοι, χαιρόμαστε που είστε εσείς ε, στο βήμα και σε αυτή τη θέση ε, και πραγματικά ε, με όλη σας την καρδιά δείχνετε ότι θέλετε να αφαιρωθείτε σε αυτήν την στρατηγική γιατί είναι πράγματι είμαστε εταίροι με την Αφρική και μοιραζόμαστε το ίδιο πεπρωμένο και από κοινού θα πρέπει να πετύχουμε. Αλλιώς θα αποτύχουμε και οι δύο πλευρές. Και αυτή είναι η πρώτη συνέπεια μια ισότιμης εταιρικής σχέσης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουν χώρο ε, βραχυπρόθεσμα εθνικά αλλά ούτε και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια εταιρική σχέση ε, για την εκπαίδευση, να αφήσουμε τα κορίτσια να σπουδάσουν, ε, ιδίω τα κορίτσια, για 10 χρόνια τουλάχιστον. Επίση, θέλουμε υγειονομική περίθαλψη, κεντρική περίθαλψη για όλου και καλέ θέσει εργασία. Όχι employability, απασχολησιμότητα. Θέλουμε καλέ θέσει εργασία για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη κοινωνία. Το ίδιο ισχύει για την Ευρώπη, το ίδιο ισχύει για την Αφρική. Αυτή είναι η δουλειά μα ε, και θα συνεισφέρουμε και εμείς και θα σας στηρίξουμε στεναρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τώρα εκ μέρου ε, τη ομάδα Ρινιού. Το λόγο έχει ο Σαρλ Γκέρενς. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Κογκό είναι η μεγαλύτερη γαλλόφωνη χώρα στον κόσμο και ανάμεσα στις χώρες που μιλούνται στην Αφρική είναι τα πορτογαλικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώς ο μεγαλύτερος εταίρος μας εμπορικός αλλά και στον τομέα της ανάπτυξης. Εννοείται ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουμε ήδη ε, προνομιακές ε, σχέσεις και ιδιαίτερα στενές. Οπότε το status quo κινδυνεύει να αποδειχτεί ιδιαίτερα αντιπαραγωγικό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια συνολική στρατηγική που να καλύπτει του τομεί, ε, το πολιτικό, τη ασφάλεια, ανάπτυξη, οικονομικό και εμπορικό. Μια πραγματική στρατηγική αυτού του μεγέθου θα πρέπει να έχει και συγκεκριμένου στόχου στον χρόνο και έναν χάρτη πορεία. Στην πραγματικότητα, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να επαναφέρουμε τη μέθοδο Ντελόρο της δεκαετίας του 90 που επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει σημαντική πρόοδο στις σχέσεις της με την Αφρικανική Ήπειρο. Σήμερα η ανάπτυξη στην Αφρική εξαρτάται ε, προφανώς από τους ίδιους τους Αφρικανούς, αλλά επίσης όλο και περισσότερο από την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία, που φτιάχνουν όλο και πιο στενούς ε, δεσμούς και σχέσεις στον οικονομικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό τομέα. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει και εμείς να δούμε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκή Ένωσης με την Αφρική. Γιατί να μην σκεφτούμε μια κοινή προσέγγιση στα θέματα της ασφάλειας και να επιτρέψουμε στην Αφρικανική Ένωση να εδρεύει στο Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ. Γιατί να μην σκεφτούμε ήδη ένα κοινό διάβημα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τι περιμένουμε για να δρομολογήσουμε μια εμπορική συνεργασία που να έχει σαν στόχο να δημιουργηθεί μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Η Αφρική πρέπει βέβαια να αναπτυχθεί η ίδια, αλλά εννοείται ότι αυτό δεν αποκλεί να έχουμε κοινέ εμπειρίε, κοινή πραγματογνωμοσύνη και κοινέ αξίε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη ομάδα ID, η κυρία Μπίλντε έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι τυχαίο αν γύρω από το Brexit, μετά το Brexit στις 20 Ιανουαρίου, το Λονδίνο ξεκίνησε τη Σύνοδο Κορυφή Αφρική Ηνωμένο Βασίλειο. Με πρωτοβουλία που μα υπενθυμίζει σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει ακόμα έδαφο στερουμένη από τον Βρετανό ε, σύμμαχο, που είναι σημαντικό παράγον διπλωματικό και εμπορικό στην Ήπειρο. Πολλαπλασιάζονται αυτέ οι σύνοδοι κορυφή. Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία. Ε, την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργό του Καναδά, ο κ. Τριντό, έκανε περιοδία στην Αφρική. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις ε, ισοτήμων σχέσεων με την Αφρική. Υπάρχουν όμως άνισες ε, αληφτικές συμφωνίες που δημιουργούν παρεμβολές ε, πολιτικές και δεν δημιουργούν κατάλληλα αποτελέσματα πολιτικά και εμπορικά. Και όσον αφορά το μεταστατικό δεν κάνουμε πολλά που είναι κρίσιμο πρόβλημα για πολλούς Ευρωπαίους. Το φορικό ερώτημα ζητούσε να επεκταθεί το έρασμος, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι θα ανοίξουμε νέες διαδρομές αφρικανικής μετανάστευσης. Η Ένωση ετοιμάζεται να επανεξετάσει την αποτυχία του Κοτονού με μια δεκαετία που έχει χαθεί. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εκ μέρους των Πρασίνων ο λόγος πάει στην κυρία Χετσμπέργκερ Φοφάνα. Η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική εδράζεται επί μια στρατηγική κοινή που παγραμμίζει τη νέα συνεργασία σε θέματα πολιτικών βάσει αξιών υποδιαπραγμάτευση κοινών ισοτήμων αξιών που καθορίζουν αυτέ τι σχέσει. Οι νέε συμφωνίε όσον αφορά αυτή τη στρατηγική συνήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ενώση, Αφρική στο Αμπιτζάν το 2017 από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που τόνισαν ιδιαίτερα τι προτεραιότητέ του ενετόπισαν τέσσερι προτεραιότητε κοινή δράση για τι επενδύσει, για το ανθρώπινο κεφάλαιο, για την αντοχή, για την ειρήνη, την ορθή διακυβέρνηση, καθώ και τι επενδύσει σε δομέ για ανάπτυξη βιώσιμη και για τη μετανάστευση. Όσον αφορά λοιπόν τη συνεργασία, ε, μέσω τη συνεργασία πρέπει να πούμε ότι αποστασιόμεθα από τι πανταλιστικέ σχέσει που επικρατούσαν μέχρι τώρα. Οι διαπραγματεύσει αφορούν τι οικονομικέ και αναπτυξιακέ σχέσει σε αυτέ τι διαπραγματεύσει προσθέτουμε και τη νέα πτυχή τη ε, στρατηγική. Αυτή η νέα πρωτοβουλία που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει πολυάριθμα ερωτηματικά όμω. Πώ μπορούμε να κρυζώσουμε την φτώχεια, πώ μπορούμε θα πετύχουμε να σταματήσουμε τι μάστιγε που φρενάρουν την ανάπτυξη για να δώσουμε προοπτικές στις γυναίκε και στους νέου σε αυτή την Ήπειρο που αποτελεί το 60% του πληθυσμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρου τώρα του ECR το λόγο έχει η κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα, κυρία Επίτροπε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΚΕ, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσεις, τη μετανάστευση. Οι νέοι που φεύγουν από την Αφρική και από άλλε χώρε ΑΚΕ και μεταναστεύουν επειδή έχουν πολύ μικρέ δυνατότητε πρόσβαση στην ε, ε, μόρφωση, σε μια αξιοπρεπή ζωή. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε και να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Αυτοί οι νέοι από τις χώρες ΑΚΕ τι χρειάζονται πάνω απ' όλα. Καλή εκπαίδευση. Η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι στην εκπαίδευση. Και πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ακριβώς αυτό το οποίο όταν δεν υπάρχει δεν επιτρέπει και την πρόσβαση στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση. Να βάλουμε λεφτά λοιπόν στην εκπαίδευση. Να επιτρέψουμε στους νέους να έχουν πρόσβαση σε μικροδάνεια και Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εγκαθιδρύσει απλούς μηχανισμούς που να επιτρέπουν στους νέους να δημιουργούν τη δικιά τους επιχείρηση στις χώρες τους, γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον πλούτο της χώρας τους. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα στρατηγική για την Αφρική. Το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται πως η Ευρώπη θέλει μια στρατηγική που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των πολιεθνικών και όχι στους στόχους ανάπτυξης και στα συμφέροντα των ε, περισσότερων Αφρικανών. Και γιατί, μην ξεγελιόμαστε, μετανάστευση, ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, όλα αυτά είναι οι γεωπολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν που χρειάζονται η Ευρώπη και η Αφρική είναι μια σχέση διάρκεια που να βασίσει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη βιωσιμότητα, στην προστασία του περιβάλλοντο. Γι' αυτό και τέτοιε στρατηγικέ δεν μπορεί να αποτελούν εργαλείο που να εξυπηρετούν τα εμπορικά ε, συμφέροντα ή τα συμφέροντα ασφάλεια τη Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε 180 μοίρε στροφή στι πολιτικέ μα για να είμαστε συνεπεί και να ε, επικεντρωνόμαστε στα δικαιώματα και συγκεκριμένα για την Αφρική δίκαιο εμπόριο, ε, νόμιμη οδή μετανάστευσης και να απαιτούμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να τηρούν τις υποχρεώσεις